Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν προβλήματα με τι μεταφορέ τη Βρυξέλλε σήμερα. Νομίζω παρόλα αυτά ότι θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, διότι τρέχει ο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξή μα. Να σα θυμίσω καταρχά ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Και πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Ε, Δυστυχώ έχουμε τροποποίησει ε, στην ημερήσια διάταξη διότι συμπίπτουν με τη συνεδρίασή μας και άλλες συνεδριάσεις. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να προτείνω να αλλάξουμε την ε, συνεδρίαση των συντονιστών και να πραγματοποιηθεί από τις 2 και 4 μέχρι τις 3 το απόγευμα. Κατόπιν έχουμε την έκθεση του Πάολο Ράντζελ που θα συζητηθεί γύρω στις 10. Και ο κύριος Μόρτεν Μέσερσμιτ συμφώνησε να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, αμέσως μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις από μένα. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Μέσο Σμιτ ε, τώρα, τον Παύλο Ραντζέλ στις 10 και την συνεδρία των συντονιστών στις 2 και 4. Η γραμματεία είναι πολύ ευέλικτη και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε τελευταία στιγμή στα αιτήματά σας. Ε, νομίζω όμως ότι υπερβάλλουμε λίγο όσον αφορά τα αιτήματα. Νομίζω ότι έχουμε υπερβολικά πολλά. Θα αναγκαστούμε λοιπόν να είμαστε πιο αυστηροί από εδώ και μπρος όσον αφορά τις ε, τροποποίηση τη ημερήσιας διάταξη στην τελευταία στιγμή. Σα παρακαλώ λοιπόν να ε, κοιτάτε την ημερήσια διάταξη όταν σα τη στέλνουμε για να αποφεύγουμε τι τροποποίησεις τη τελευταία στιγμή, διότι έχουμε παράπονα από του άλλου συναδέλφους ε, σχετικά με τι πολλέ τροποποίησει. Αυτά όσον αφορά τις τροποποίησεις της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις ή επιθυμίες για περαιτέρω τροποποίηση, ε, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη όπως διαταξη όπω εγκριθηκε Όσον αφορά το δεύτερο σημείο της ημερησίας διάταξης, ανακοινώσεις της Προέδρου, δύο ανακοινώσεις. Έχουμε παράταση της προθεσμίας ε, για τροπολογίες για την ε, έκθεση του Γκί Φερχόφστατ. Η νέα προθεσμία είναι 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι. 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι είναι η νέα ε, προθεσμία για τις τροπολογίες ε, για την έκθεση του Γκί Φερχόφστατ σχετικά με τις πιθανές ε, εξελίξεις ε, και προσαρμογές όσον αφορά την θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουμε την εισηγήτρια για την πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η Κλάουντια Ταπαρντέλ θα είναι η συγκήτρια από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και θα ήθελα τώρα να προχωρήσω στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, ε, που είναι η γνωμοδότηση του Μόρτεν Μέσερ Σμιτ για την έκθεση πρωτοβουλίας ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Μόρτεν, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ευελιξία που επιδεικνύεται δεδομένων των δυσκολιών που προκύπτουν. Όπως βλέπετε στο σημείο 10, έχουμε μία έκθεση του συναδέλφου Ντεγιόν που επισημαίνει κάποιες από τις ελλείψεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα, ε, είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλους οργανισμούς όπως είναι ο και άλλοι από τον Ιανουάριο του 2014 είναι υποχρεωτικό για τα θεσμικά όργανα να έχουν διαμορφώσει πολιτική για την ε, προστασία των ε, μαρτύρων ε, δημοσίου συμφέροντος. Σίγουρα λοιπόν είναι ώρα να κάνουμε κάτι. Έχουμε λοιπόν την γνωμοδότηση σε 8 σημεία δεδομένων των περιορισμών. Προσπαθώ να τονίσω τα σημαντικά. Λέω μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συγκεκριμένο κεφάλαιο για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, τις καταγγελίες για διαφθορά και απάτη. Αυτό είναι απαραίτητο, γι' αυτό το έχω συμπεριλάβει αυτό στο σημείο 7 και όπως λέω στο σημείο 8 ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, ενθαρρύνσεις της διαμεσολαβήτριας ε, να υπάρχει σαφής ε, διάκριση ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς ε, κάνουν ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη. με κάποιου περιορισμού ε, που δεν ενδιαφέρουν για την μας ε, επιτροπή. Νομίζω ότι η έκθεση του κ. Ντελιών είναι πολύ καλή, ε, είναι φιλόδοξη, έχει τη σωστή προσέγγιση και γι' αυτό έχω περιορίσει τη δική μου γνωμοδότηση στο να επισημαίνω κάποια σημαντικά στοιχεία και έχω περιοριστεί σε κάποιες μικρές προσθήκες. Ε, πάντως προσβλέπω στην συζήτηση σήμερα με τους ε, συναδέρφους. Ε, ευχαριστώ σας συζητήσουμε τις τροπολογίες σας και ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλει κανείς να μιλήσει εκ μέρους της Περβάνς Περές από τους σοσιαλιστές. Ρίτσαρντ, όχι όμως ως και ο Τότε σε παρακαλώ να περιμένεις λίγο να ακούσουμε πρώτα τους εσκιώδεις εισηγητές. Ε, ο κ. Ιαντός και η Σιλβί Κουλάρ ή κάποιος άλλος. Σιλβί Κουλάρ από την Άλτε, δεν έχουμε κανέναν παρόντα. Μπάρμπαρα Σπινέλη από την ΚΟΕ, ούτε βρίσκεται εδώ κανείς άλλος να μιλήσει. Ο Μαξάντερσον είναι εδώ όμως. Ε, μήπως θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ ως κοιόδης εισηγητής. Οι οικολόγοι πράσινοι πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας πάνω στο θέμα αυτό. Δεν έχω προετοιμαστεί, κυρία Πρόεδρε, για μια τέτοια παρέμβαση. Περιμέναμε άλλωστε να συζητηθεί αργότερα το θέμα αυτό. Πάντως, σε γενικές η, η ε, γνωμοδότηση αυτή ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση και προσβλέπουμε στην ε, ε, συνέχιση της δουλειάς. Πρόεδρος, αυτό ακριβώς δείχνει τις συνέπειες των τροποποίησεων τελευταίας στιγμής της ημέρησιας διάταξης, ότι δεν έχουμε συναδέλφους προετοιμασμένους για τη συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν να περιοριστούν αυτές οι τροποποίησεις στο μέλλον. θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιες ερωτήσεις έχω. Καταρχάς, στο τρίτο σημείο του σχεδίου γνωμοδότησης ε, λέει ότι εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από όλα τα θεσμικά όργανα και όλους τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που συνάδει με το σημείο 9 του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Ντεγιόν που καλεί όλα τα θεσμικά όργανα που δεν το έχουν ήδη κάνει να εφαρμόσουν το άρθρο 22 γάμα ε, του ε, κανονισμού. Ποια θεσμικά όργανα δεν το έχουν κάνει ακόμα. Θα ήθελα αυτό να λέμε αντί απλά να λέμε ότι να το κάνουν όσοι δεν το έχουν κάνει. Αν ε, λοιπόν ε, έρθετε σε επαφή με τον κύριο Ντεγιόν, θα ε, πρότεινα να του το πείτε αυτό, να μην κάνουμε μια γενική παρατήρηση, να λέμε συγκεκριμένα ποιο δεν το έχει κάνει. Και όσον αφορά το σημείο 8 του σχεδίου γνωμοδότησή σα, λέει καλή την Επιτροπή να επιληφθεί το αιτήματο τη διαμεσολαβήτρια. Δεν βλέπω όμω πουθενά τι είναι το αίτημα τη διαμεσολαβήτρια. Ούτε το δικό σας κείμενο, ούτε με μια γρήγορη ανάγνωση το βρίσκω στο κείμενο του κύριου Ντεγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελες να μιλήσεις ε, εκ μέρους της Κωνσταντσε ή δικές σου παρατηρήσεις έχεις. Δικές μου παρατηρήσεις έχω, κυρία Πρόεδρε. Θα συμφωνούσα με τον Ρίσαρτ ότι η αλλαγές στην ημερήσια διάταξη ε, έχουν κάποιες ε, απρόβλεπτες συνέπειες. Όσον αφορά τους ε, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ας είναι σαφές ότι είναι πολύ χρήσιμος ο ρόλος τους και ο στόχος τους. Και νομίζω ότι μιλώ και στο όνομα του συνόλου του ΕΛΚ στο θέμα αυτό. Δεν έχω ακριβώ επιφυλάξει. Έχω ερωτήσεις σχετικά με την όλη ιδέα. Νομίζω ότι είναι σχετικά νέα η ιδέα. Οποιοςδήποτε όμως προέρχεται από κομμουνιστική ε, χώρα δεν θα μπορεί να κάνει τη διάκριση ανάμεσα ε, σε έναν πληροφοριοδότη της αστυνομίας ε, και έναν μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Προσπαθούμε να πούμε ότι είναι καλό να λέτε ε, να καταγγέλλετε τους εργοδότες σας αν πιστεύετε ότι κάνουν κάτι λάθος. Ε, μπορεί αυτό να είναι απόλυτα σοφές, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει η διάκριση ε, ανάμεσα στους ε, άτυπους πληροφοριοδότες, για παράδειγμα, στην Ανατολική Γερμανία και τους ε, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που έχουμε εδώ πέρα. Ποια λοιπόν είναι τα εχέγγυα ώστε να αποφύγουμε ε, τους μάρτυρες, ε, ε, τους κακόβουλους. Κάτι που είναι δύσκολο να αποφύγουμε. Τι χέγγια λοιπόν έχουμε για να μην τεινάξουμε όλο το σύστημα στον αέρα. Έχουμε εδώ πέρα τεκμήριο αθωότητας. Έρχεται ο κύριος Χ και λέει για την κυρία Ψ ότι κάνει κάτι περίεργο με τα χρήματα. Υπάρχει όμως το τεκμήριο αθωότητας και δεν ε, θα πρέπει να θεωρείται απόλυτη αλήθεια αυτό που λέει ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, ε, ενώ είναι αρκετά σαφής ο τίτλος ότι μιλάμε για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ε, πού τελειώνουν τα οικονομικά συμφέροντα και πού ξεκινάνε θέματα εξουσίας. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πρόεδρε, εσεί και οι άλλοι από πρώην κομμουνιστικέ χώρες θα γνωρίζουν ότι το να ενθαρρύνουμε ε, τέτοιε καταγγελίε ε, οδηγεί ε, σε σε πολλές επιφυλάξεις στους ανθρώπους, δηλαδή προτιμούν να είναι πάντα ασφαλείς. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαίνει ότι σε μια δημοκρατία μεγάλου μεγέθους Ε, είναι πολύ δύσκολο να χειριστεί κανείς τέτοια θέματα ε, και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ε, μια ερώτηση. Πού σταματάει η καταγγελία δυσλειτουργιών και πού ξεκινάει και πού ξεκινάνε οι κακόβουλες καταγγελίες. Ευχαριστώ. Η Mercedes Ευχαριστώ, Πρόεδρε. συμπαθάτε με, αλλά ο Ραμόν αργη που είναι ο σκιώδης ε, εισηγητής μας ε, θεώρησε ότι θα τα συζητήσουμε το απόγευμα. Τέλος πάντων μου έδωσε αυτό το σημείωμα. Θα το δώσουμε στον ε, εισηγητή σε αυτό το σημείο λέει ότι είναι υπέρ του βασικού κειμένου. Και λέει ότι υπάρχει το πρόβλημα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Όσον αφορά την ε, καταγγελία ε, των ε, απατών, την καταγγελία τη σχετική με κάποιες αθέμητες πρακτικές. Οπότε, με δεδομένα αυτά το πει ο κύριος ε, Σέφλιν, θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί του. Εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε κάποιου είδους ε, καταγγελίες οι οποίες να είναι θέμα κυρίως εθνικής πολιτικής. Αφορώντας φυσικά κάποιες ε, ε, αθέμητες πρακτικές, κάποιες απάτες. Επότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συγκροτήσουμε μια υπηρεσία που να αξιολογεί το κατά πόσο ευσταθούν οι σχετικές ε, καταγγελίες. Γιατί βέβαια πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος της συκοφαντίας. Άρα, ποιος καταγγέλει, πώς στοιχειοθετείται το καταγγελόμενο και επίσης να δούμε πώς θα πλαισιώσουμε αυτόν τον μηχανισμό που έχει σχέση με την ε, καταγγελία. Μπορεί δηλαδή κάποιος να μην έχει κάνει καμία θεμετή πρακτική και να συκοφαντείται. Είναι πραγματικό το πρόβλημα. Βέβαια το, το λεπτό ζήτημα εδώ είναι ότι αυτό είναι θέμα ίσως και αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ. Μπορεί να υπάρξει συσκομφαντία και κατά φυσικού προσώπου και κατά ε, θεσμικού οργάνου. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό, να το μελετήσουμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που έχουμε και να δούμε το πώς θα ελέγχουμε το τι ισχύει για αυτόν ο οποίος προέβησε μια καταγγελία. Προσοχή επομένως όσον αφορά τον ενθουσιασμό για κάτι το οποίο προέκυψε. Να βλέπουμε πάντοτε αν υπάρχει τεκμηρίωση. Να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό του ότι ανακαλύφθηκε δηλαδή κάποια μεγάλη απάτη οικονομική γενικότερα. Να μην φτάσουμε σε καταστάσεις δικτατορικών καθεστώτων όπου εκεί πέρα πάρα πολύ εύκολα ε, και αβίαστα κανείς καταλήγει σε κατηγορίες και καταγγελίες. Προσεγγιμένως να περιφρουρήσουμε την φήμη, το όνομα προσώπων ε, ε, από τέτοιες καταγγελίες, τέτοια φαινόμενα. Thank you very much. Anybody else would like to... Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. άλλος τον λόγο. ή Ιδάλλως Πεςτε μας. Σας ευχαριστώ για όσα είπατε και ήθελα να πω πρώτα πρώτα προς την Mercedes ότι όλοι συμφωνούμε. Αυτά λέει και ο Τζόρτζ. Η προστασία των καταγγελόντων από την άλλη μεριά να περιφρουρήσουμε την αρχή του τεκμηρίου αθωότητος να μην υπάρχει κακόβουλη χρήση της καταγγελίας άλλωστε αποτελεί έγκλημα το να καταγγείλει κανείς κάτι γνωρίζοντας ότι η κατηγορία δεν είναι αληθής. Άρα, ελεγκτικός μηχανισμός. Επομένως να υπάρξει κάποια υπηρεσία που να αξιολογεί Α, και η Όλαφ θα μπορούσε να συνεργαστεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε την Όλαφ, γιατί να φτιάξουμε καινούργια υπηρεσία. Θα μπορούσε αυτό να συζητηθεί και στη ΛΥΜΠΕ, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και αλλού. Κύριε Κόρμπετ, καλά τα είπατε. Όντω, ε, στα σχετικά σημεία ε, δεν κατάφερα να τα πω κρυστάλλινα. Ε, έχετε δίκιο, συμπαθάτε με. Υπάρχει εδώ πέρα θεσμικό έλλειμμα και επίσης θα πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα του διαμεσολαβητή σε σχέση με την ετήσια έκθεσή του και αυτά τα όσα ζητεί, προτείνει κλπ. Να διευκρινιστούν αυτά τα σημεία. Και έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα που δεν είναι τόσο πολιτικού χαρακτήρα, είναι πιο πολύ ακαδημαϊκού, φιλοσοφικού. Συνεχίσουμε το συζητούμε. Σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Thank Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι στις δύο έκτακτες επιτροπές για τις φορολογικές συμφωνίες συζητήθηκε το ζήτημα των καταγγελόντων. Όλα αυτά αναφέρονται και στις σχετικές εκθέσεις. Για να δούμε τώρα τις τροπολογίες. Οι προθεσμίες 5 Οκτωβρίου, σημαντική ημερομηνία. 5 Δεκάτου το μεσημέρι. Όχι. 6. 6 ώρα το απόγευμα. 6 μετά μεσημβρία της 5ης Οκτωβρίου. of 6 p.m. Uh, μεσημβρία στις 5 Δεκάτου και θα ψηφίσουμε στη δεύτερη συνεδρίαση στις 20 Οκτωβρίου και 8 ενδεκάτου η τελική ψηφοφορία δεν θα δοθεί παράταση της τροπολογίας γιατί δεν θα προλάβουμε έτσι να τηρήσουμε την προθεσμία την τελική ψηφοφορία. Το τελειώσαμε αυτό στην μέση διάταξη. Και... It's a bad one uh, because we have half an hour till Mr. Paolo Rangel comes and Mr. Ujazdowski is prepared to make his presentation. Ε, θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Ράντζελ για να έχει να παρουσιάσει τη δική του νομοδότηση. Οπότε θα περάσουμε ε, στην. Ε, προτείνω να περάσουμε στην εξέταση της ε, του κυρίου Γιαντόφσκι, αν συμφωνείτε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει, Εάν όχι, αυτό θα κάνουμε. Θα περάσουμε δηλαδή απευθεία στην εξέταση τη ε, γνωμοδότησης του κ. Ζαντόφσκι. Έχετε το λόγο. Έχεις, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μου γνωμοδότηση αφορά λοιπόν το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες και πρόκειται για μια γνωμοδότηση η οποία ε, καταρτίζεται από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία και κατά συνέπεια εμεί συντάσσουμε από τη δική μα πλευρά κάποιε συστάσει σε ό,τι αφορά το μέλλον του λόγου προγράμματο. Θα θέλαμε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στο λόγο πρόγραμμα και θέλουμε οι αιτήσει στόχοι του λόγω προγράμματος να είναι πολύ σαφείς. Εκείνο που επίσης ε, επιθυμούμε, ζητούμε, είναι να υπάρχει, να υιοθετήσουν ένα πιο ανοιχτό χαρακτήρα τα εθνικά σημεία επαφής και ζητούμε επίσης να προωθηθεί πιο εντατικά ε, στα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατομελών το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Με άλλα λόγια θέλουμε να δώσουμε το έναυσμα στα μέσα ενημέρωσης να ε, δώσουν περισσότερη προβολή ε, σε αυτό το πρόγραμμα και τέλος η δική μου γνωμοδότηση ε, προτείνει την ανταλλαγή εμπειριών ε, μεταξύ του Εράσμους, της Δημιουργικής Ευρώπης και αυτού του, του προγράμματος της Ευρώπης για τους Προτείνουμε επίση την ανταλλαγή εμπειριών αλλά και βέλτιση των πρακτικών μεταξύ του προγράμματος μας, δηλαδή του προγράμματο Ευρώπη για τους πολίτες και του, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ε, Πολιτών. Και αυτό γιατί και τα δύο αυτά προγράμματα στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής ε, στα κοινά των πολιτών. Μία ακόμα σύσταση που κάνουμε αφορά ε, τα προγράμματα εκείνα, τα project δηλαδή, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι αρχές λοιπόν που είναι αρμόδιες για την έγκριση των ε, project, στα πλαίσια του προγράμματος, θεωρούμε ότι όταν ε, αποφασίζουν να απορρίψουν μια υποψηφιότητα θα πρέπει να εξηγούν με σαφήνεια τους λόγους της απορρίψης στους ενδιαφερόμενους, στους υποβάλλοντες δηλαδή, την λογοπρόταση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η αξιοπιστία του συνολικού προγράμματος. Και τέλος, προτείνω να ανοίξει εντός εισαγωγικών περισσότερο το πρόγραμμα, δηλαδή να καταστεί προσβάσιμο σε ε, χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, στοχεύουμε βέβαια κατά κύριο λόγο στις μη κυβερνητικές οργανώσεις των εν λόγω υποψηφίων χωρών. Αυτά σε γενικές ε, γραμμές περιλαμβάνει ως περιεχόμενο η νομοδότηση, αλλά όπως είπα η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Οι δικές μας ε, συστάσεις ε, προφανώς θα πρέπει να αφορούν την εντολή της δικής, της δικής μας ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και ακριβώς με αυτό το σκεπτικό συνέταξα το κείμενο της νομοδοτησής μου. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πάρει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ, γιατί βλέπω ότι είσαι ο μόνος από την πλευρά της πολιτικής ομάδας. Ναι. Ε, από την πλευρά μου, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ζαντόφσκι για αυτήν την ε, παρουσίαση της γνωμοδότηση. Ένα σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να θέσω εδώ και θα μπορούσα να το θέσω και ω ερώτημα είναι το εξή. Ε, προωθούμε την έννοια της ηθαγένειας του citizenship σε, ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το πρόγραμμα ή όχι, γιατί έχει εκφραστεί εκτεταμένη αμφισβήτηση ε, για παράδειγμα ε, στη δική μου χώρα στην ε, Ουγγαρία δηλαδή έχουμε ήδη την ηθαγένεια της Ουγγαρίας τι σημαίνει το να έχουμε ευρωπαϊκή ηθαγένεια και άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα αυτά της περιαγωγής και άλλων μπορούν να συμβάλλουν ακριβώς στην οικοδόμηση μιας τέτοιας έννοιας ηθαγένεια, στην καλύτερη κατανόησή της και σε ευρύτερη κλίμακα. θεωρώ πως είναι καλή ιδέα το να θέλουμε να επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα σε υποψήφιε χώρε ε, και όχι μόνο στι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά και ακόμα ε, πιο ευρέω. Και ε, η αναφορά που κάνετε σε ό,τι αφορά το Εράσμου είναι μία από τι πλέον χρήσιμε. Νομίζω πως όλοι συμφωνούν ότι το Εράσμος αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ό,τι διαβάζω ε, στο Βρετανικό ε, τύπο υπάρχει πραγματικά μεγάλη απελπισία για το γεγονός ότι ενδεχομένω ε, χιλιάδες εφηρητών και νέων μπορεί να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στο Εράσμους ενώ είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν μέχρι τώρα να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Οπότε πραγματικά έχει αξία αυτή η αναφορά που κάνετε στο Εράσμους. Τώρα δεν ξέρω την να πω σε σχέση με αυτήν την αναφορά που κάνατε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Γνωρίζετε πως εγώ είμαι υπέρ αυτής της ε, πρωτοβουλίας ουσιαστικά υπνοβατή, δηλαδή βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Επιτροπή και να τη ρωτήσουμε τι κάνει. Ίσως ε, ε, όταν θα καλέσουμε και πάλι τον κύριο Τίμερμαν να έρθει εδώ στην Επιτροπή μα, ίσως τότε θα πρέπει να του θέσουμε το σχετικό ερώτημα σχέση με το τι συμβαίνει με την Πρωτοβουλία. Αυτά ε, από τη δική μου πλευρά ε, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη γνωμοδότηση, αλλά σε κάποια σημεία, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ακριβώ το πρώτο που έθεσα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εδραίωση τη ίδια ε, τη Ευρωπαϊκή Ιταγένεια, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να προβούμε σε κάποιε βελτιώσει τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, Τζορτζ Μαρσέλα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Και εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί έχουμε αυτές όλε τι αλλαγέ στην μέση διάταξη. Αλλά τέλος πάντων. Ε, δυσκολήθηκαν πράγματα για να συνηθούμε με τους σκιώδες τους άλλους. Οπότε, τι να σας πω τελικά, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, γιατί α, προηγουμένως τοποθετήθηκα από τη βάση των όσων μου είπαν οι συνάδελφοι, αλλά τώρα προσωπικό λέμε. Ε, οπότε, με αυτά που άκουσα από τους συναδέλφους ε, ε, είμαι πεπισμένη ότι τώρα διαμορφώνεται ακριβώς αυτή η ιδιότητα του Ευρωπαίου του Ευρωπαίου πολίτη και βέβαια ανά κράτος μέλος ποικίλει το ενδιαφέρον, η συνειδητοποίηση σε σχέση με τη γνώμη για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς το πόσο κανείς είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί με το θέμα. Και έχουμε αυτή την επίσκεψη του Ελβετού πρέσβεως που είπε ότι ακριβώς αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα μετά από κάποια αποστολή στην Ιαπωνία. Αυτό το αίσθημα του ανήκει δηλαδή στην, ε, στην Ευρώπη. Βεβαίω και έχει σημασία το έρασμος. Είναι θέμα της κινητικότητας στην Ευρώπη των Ευρωπαίων. Μια συγκεκριμένη εμπειρία Ακριβώς όταν κάποιος εγκαταλείπει την ε, Ευρώπη, τότε συνειδητοποιεί τι πάει να πει το να έχουμε κοινά θεσμικά όργανα, κοινούς κανόνες, για την οικονομία, για το περιβάλλον, ε, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο, το θέμα των ε, δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην Ευρώπη. Τότε ακριβώς νιώθει τι πάνε να πούν όλα αυτά. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν τους νέους σχετικά. Σε σχέση με αυτή τη, την συνάντηση που αφορά τους νέους, αυτή τη διάσκεψη τέλο πάντων, για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων τους και των Ευρωπαίων γενικότερα την ε, ελεύθερη διακίνηση των προσώπων να, τι τονώνει το αίσθημα αυτό του ανήκει στην Ευρώπη. Αυτές οι πρωτοβουλίες αλλά ότι είναι, δεν είναι νομοθετικό χαρακτήρα, Προκειμένου για κάποιες δραστηριότητες, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη γνώση της Ευρώπης, των δικαιωμάτων, όλα αυτά που με θετικό τρόπο ορίζουν το τι πάει να πει Ευρώπη. Και βέβαια θα πρέπει να γίνει και αξιολόγηση ότι πρέπει να μεταβληθεί από αυτό το προστάσιο. Και άρα στην επιλογή μας, στην απόφασή μας θα πρέπει να λαμβάνετε απόψη το σε ποια κοινωνική ομάδα στοχεύουμε κάθε φορά με μια πρωτοβουλία. Πάντως βασικά μιλούμε για τις νέες γενιές. Υπάρχουν αυτά τα δίκτυα σχολείων, ε, νεολαίστικων οργανώσεων, να, που θα δώσουμε την προτεραιότητα. Οι νέοι είναι αυτοί που θα πρέπει να προβληματιστούν, ε, να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους, κάτι που θα κρίνει και το μέλλον τους και αυτοί τελικά θα επιφέρουν τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν, δεν είναι παθητική η γνώση που αποκτά κανείς με αυτά τα προγράμματα. Ε, εκεί κανείς συμμετέχει ενεργά και μαθαίνει. Έτσι μεταλαμπαδεύεται λοιπόν το φεντρελιστικό ομοσπονδιακό πνεύμα. Και φυσικά δεν έρχεται σε αντίφαση όλη αυτή η προσπάθεια του ανήκειν στην Ευρώπη με την, το, το, το ανήκειν στην κοινότητα, από όπου προέρχεται ο καθένας, την πιο μικρή. Πολύ σημαντικά αυτό. Τώρα, τέλος έχω να σας πω ότι συμφωνώ στα υπόλοιπα, όπου δεν συμφωνώ θα έχουμε, κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες. Είναι σημαντικό λέγω ότι θα, θα πρέπει να δούμε το ότι θα πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες να επεκταθούν και στα νέα, στα υποψήφια για ένταξη κράτη, στα κράτη επίση που έχουν συμφωνίε σύνδεση. Άρα, όλη αυτή η προβληματική να ξεπεράσει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να έχουμε ε, αυτού του είδου την ε, εμπλοκή των ε, νέων, την επαφή μεταξύ νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων εκείνων των χωρών και έτσι ακριβώς να αισθανθεί ο κόσμος ότι πάει να πει το ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Και σας παραπέμπω στο έκτο σημείο του κειμένου που νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε για το έργο σας κύριε Ισηγητά και η συντονίστριά μας θα συμβάλλει όσο μπορεί. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, μιλήτρια, όχι συντονίστρια, η σκιώδηση εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας. Θα ήθελε κανείς να μιλήσει από την Άλτε, ούτε από την Κούα έχουμε κανέναν. Οι πράσινοι δεν έχουν ορίσει σκιώδη εισηγητή. Μαξ Άντερσον, παρακαλώ. Δεν μιλώ στο όνομα της ομάδας, διότι η πολιτική μας ομάδα έχει πολύ πιο ε, θετική άποψη για το πρόγραμμα αυτό από ό,τι έχω εγώ. έχω κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με το αν αυτό αποτελεί καλή χρήση χρημάτων, εάν θα είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Υπάρχει μήπως στοιχείο προπαγάνδας στο πρόγραμμα αυτό. Δεν αποτελεί προτεραιότητά μου το θέμα αυτό. Προσέχω όμως ότι φαίνεται να δίδεται διαφορετική έμφαση στη γνωμοδότηση από ό,τι στο πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό. Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, να ρωτήσω τον κύριο Ουιαστόφσκι αν θα ήθελε να ξαναμιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας. Θα αναφερθώ πρώτα στην τελευταία παρέμβαση. Μήπως δηλαδή υπάρχει κίνδυνος ε, το πρόγραμμα αυτό να εξυπηρετεί στόχους αποκλειστικά προπαγανδιστικούς. Η γνωμοδότησή μου προσπαθεί ακριβώς να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αυτόν. Ζητάμε καλύτερο ορισμό των στόχων και περισσότερη διαφάνεια στο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ αξιολογώ θετικά το πρόγραμμα και έχω διατυπώσει την γνωμοδότηση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε περαιτέρω τους στόχους του προγράμματος κατέγραψα τις παρατηρήσεις της κυρίας Πρέσο και του κυρίου Σοπφλίν. Και είμαι διατεθειμένος να εισάγω και κάποιες πτυχές που αφορούν τη νέα γενιά, ε, στην οποία απευθύνεται κυρίως το πρόγραμμα. Καθώς και να αναφερθώ στις ανταλλαγές εμπειριών και στις επαφές μεταξύ νέων. Όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή υπηκότητα, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σιωφλίν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ένα στοιχείο προφανές. η ε, εντύπωση που δόθηκε στον ε, Ελβετό πρέσβη μάλλον είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και τα επιμέρους ε, εργαλεία όπως είναι η πρωτοβουλία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι χρήσιμο να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να δημιουργηθούν δεσμοί ανάμεσα στο πρόγραμμα ε, Ευρώπη για τους πολίτες ε, με την ε, πρωτοβουλία για τους πολίτες. Και θα ήθελα να... Έπασε τόσο έχω σημειώσει τις παρατηρήσεις. Πρόεδρος, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. και να ψηφίσουμε ε, τον Νοέμβριο. Ο κύριος Ράντζελ, από ό,τι φαίνεται, ε, καταφθάνει. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να διακόψουμε. Μήπως μπορεί κάποιος ε, να μας διασκεδάσει λίγο μέχρι να καταφθάσει, διότι βρίσκεται ακόμα στην άλλη άκρη του κτηρίου. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Ράντζελ. Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε ε, με τη συνεδρίασή μας γιατί έχει προσέλθει ο συγκητής για το επόμενο θέμα. Απλώς ε, δεν ξέρω... Έχω κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση του κ. και γιατί το 2006 είχε ληφθεί μια κοινή απόφαση Ρίτσαρντ, ίσω ε, μπορεί να μα βοηθήσει εδώ να το διευκρινίσουμε. Έχει ληφθεί λοιπόν μια κοινή απόφαση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και από εκεί και μετά η επέκταση του προγράμματο το 2014 έγινε μέσω κανονισμού μόνο του Συμβουλίου, χωρί δηλαδή να έχει συναποφασίσει τον νόμο κανονισμό το Κοινοβούλιο. Μήπω ε, θα έπρεπε λοιπόν να τεθεί αυτό το ζήτημα στη γνωμοδότησή μα. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί συνέβη αυτό, γιατί η επέκταση έγινε μόνο από το Συμβούλιο. Ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο προσεκτικότερα. Καλώς σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε πλέον πραγματικά την εξέταση αυτού του σημείου. Οπότε θα ήθελα να ε, περάσουμε στο θέμα που αφορά την εφαρμογή των ε, διατάξεων της συνθήκης ε, που αφορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια με τον με μας τον Σάρφο Παύλο ε, και να σας κάνω μια εισαγωγή από την πλευρά μου έτσι πολύ σύντομη. Όπως γνωρίζετε έχει υπάρξει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τους ε, τον εσωτερικό κανονισμό και το πλαίσιο που αφορά την υποβολή των ε, εκθέσεων εφαρμογής των implementation reports, ε, οι οποίες πλέον ενθαρρύνονται από όλες τις πλευρές για υποβολή. Άλλαξαν λοιπόν οι κανόνες σε ό,τι αφορά την υποβολή αυτών των εκθέσεων εφαρμογής και στο πλαίσιο εκείνο η ΑΦΚΟ είχε προτείνει και το πεδίο που καλύπτουν αυτές οι εκθέσεις εφαρμογής να διευρυνθεί έτσι ώστε να αφορούν ε, και την εφαρμογή και την επιβολή της ίδιας της συνθήκης, κάτι δηλαδή το οποίο δεν ήταν δυνατό στο πλαίσιο των προηγούμενων ε, εκθέσεων ε, εφαρμογής. Άρα λοιπόν ε, κατά αυτόν τον τρόπο ε, η εντολή και το δικαίωμα του να συντάσσει τέτοιου είδου ε, εκθέσει εφαρμογή η Επιτροπή ΑΦΚΟ έχει διαβρινθεί Οπότε νομίζω πω και εδώ απευθύνομαι ιδιαίτερα στου συντονιστέ. Θα ήταν καλύτερο να συντάξουμε περισσότερε τέτοιε εκθέσει εφαρμογή γιατί υπάρχουν ένα, μια σειρά από ζητήματα τα οποία σχετίζονται ακριβώ με την εφαρμογή και την επιβολή τη συνθήκη και αφορούν τα ζητήματα των οποίων άπτεται η Επιτροπή μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση εφαρμογή ε, των διατάξεων που αφορούν ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα δώσω το λόγο στον συγητή του κύριο Ράντζε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που κάνατε, γιατί ε, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό το να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την ιδέα της εφαρμογής των εκθέσεων δηλαδή εφαρμογής ως ένα είδος αξιολόγησης ε, του κεκτημένου μας, του τι συμβαίνει, του status quo, που βέβαια με τη σειρά της μια τέτοια αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική για να δούμε το τι συμβαίνει, όχι μόνο στο πλαίσιο των ε, υφιστάμενων συνθήκων, αλλά και στο πλαίσιο των μελλοντικών συνθήκων που θα έχουμε. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας το γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν πλέον πολύ πιο ισχυρή παρουσία και πολύ μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτικού γίγνεσθε, ε, ειδικότερα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό βέβαια συμβαίνει για πολύ καλούς λόγους, αλλά συχνά τα κοινοβούλια αυτά ε, υιοθετούν μια πολύ επικριτική στάση, ε, όχι, αν όχι σκεπτικιστική, εν πάση περιπτώσει εκφράζουν αμφιβελίες σε ό,τι αφορά τον, το ε, ευρωπαϊκό πολιτικό κόσμο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εγώ κατονόμασα αυτή τη στάση που υιοθετούν κάποια εθνικά κοινοβούλια ένα είδος θεσμική ζήλια, αν θέλετε. Δηλαδή, η συνθήκη τη Αβώνα ε, δημιούργησε κάποιε προσδοκίε ότι θα υπήρχε με αποτέλεσμα την ε, εντατικότερη συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ τους, αλλά ότι θα υπήρχε σύγκληση στις ιδέες τους. Ως δηλαδή ε, προς ε, τον ε, εκτελεστικό ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς τον ρόλο που έχει αναλάβει το Συμβούλιο Ε, για το οποίο έχουν εφεύρει και οι Ιταλοί μας ε, φίλοι έναν ε, ξεχωριστό όρο. Κατεύθυνση. Μάλλον κατεύθυνση πολιτική. άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η προσδοκία από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων να μπορούν να συμμετέχουν και να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα την πολιτική διαδικασία στα θεσμικά όργανα. Όμω η εμπειρία που έχουμε από, τα, ε, από την ΚΟΖΑΚ, δηλαδή από τη Συνέλευση των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, ε, διαπιστώνουμε ότι, έχω διαπιστώσει εγώ προσωπικά, ότι αντιλαμβάνονται πολλά εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω ανταγωνιστή του. Και αυτό με ανησυχεί πολύ, γιατί βέβαια δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό ο σκοπό τη συνθήκη τη Λισαβόνα και αποτελεί μια λανθασμένη προσέγγιση από την πλευρά τους. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αγώνα που δίνουμε από την πλευρά μας, σε ό,τι αφορά την ε, περισσότερη νομιμοποίηση και την ε, ισχυρότερη δημοκρατικοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή η στάση των Εθνικών Κοινοβουλίων αποτελεί γεγονός όπως και ο εθνικισμός ο οποίος ε, πραγματικά χέρι υποστήριξη σε πολλά κράτη-μέλη. Κατά συνέπεια λοιπόν η στάση που έθετουν αλλά και η ρητορική ε, που υιοθετούν πολλά εθνικά κοινοβούλια είναι αρκετά εμφατική. Οπότε Ε, το ίδιο το θεσμικό ζήτημα, ε, πολιτικό θεσμικό ζήτημα, ε, δεν είναι το αμυγές αντικείμενο αυτής της γνωμοδότησης. Δηλαδή, εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να λύσουμε την κατάσταση και από εκεί και μετά να χαράξουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Αυτά εν είδη εισαγωγικών σχολείων δεν θα είμαι μακροσκελής, γιατί εκείνο που θεωρώ πως είναι πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ένα είδος brainstorming, δηλαδή να αναφέρει ο καθένας τις του ιδέες. Ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να, να, να υποβάλει εδώ τις ιδέες του ως προς ε, ε, το έργο που θα κληθώ ε, να κάνω στο πλαίσιο αυτής της νομοδότησης μέσα στους επόμενους μήνες. Και προφανώς θα πρέπει να δώσουμε και την κατάλληλη έμφαση στην, στο διερευνητικό σκέλος αυτής τη διαδικασία. Ε, δηλαδή θα πρέπει να διαπιστώσουμε πώς έχουν τα πράγματα, τι συμβαίνει επί τόπου. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε στην πράξη ποιο είναι ο βαθμός εφαρμογή αυτή τη αρκετά φιλόδοξή ε, συνθήκη των φιλόδοξων στόχων της συνθήκης της Λισαμπόνας. Η συνθήκη είναι πάρα πολύ σημαντική και κατά συνέπεια θα πρέπει να διαβουλευτούμε να συμβουλευτούμε τα Εθνικά Κοινοβούλια, εμπειρογνώμονε. θα πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία, ώστε να αξιολογήσουμε το πώς έχει κατάσταση σε ό,τι αφορά τους επιμέρους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους στα Εθνικά Κοινοβούλια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα όσα προβλέπονται στα πρωτοκολλά 1 και 2. η επιβολή η εφαρμογή στην πράξη ε, των ε, αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων των εθνικών κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πολιτικό ε, νομίζω πως ε, δημιουργεί κάποια δυσκολία ως προς το ότι δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ακριβώς τις αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές αρμοδιότητες. Ε, είναι σαφές ότι τα εθνικά κοινοβούλια επιθυμούν να ε, έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν αμυγός ευρωπαϊκά σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ακριβώς αυτός ο διαχωρισμός των εξουσιών αν θέλετε στο πλαίσιο της ε, συνθήκης της Ισλαβώνας δηλαδή το τι αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ακριβώς σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ λογική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την τήρηση των αρχών της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δηλαδή το πώς εμείς, ε, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και η Επιτροπή, το πώς λοιπόν εμείς έχουμε ερμηνεύσει τις αρχές της ε, επικορικότητας και της αναλογικότητας όπου χρειάστηκε να δοθεί μια τέτοια ε, ερμηνεία. Αυτό θα μας βοηθήσει ακριβώς να διακρίνουμε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις ε, εθνικές αρμοδιότητες, δηλαδή τις αρμοδιότητες των ε, κοντινόπουλών για τα κράτη-μέλη και τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Ε, αυτό είναι σημαντικό να γίνει και φυσικά σχετίζεται στενότατα με τις ε, διαδικασίες της κίτρινης κάρτας και της πορτοκαλί κάρτας. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πόσες φορές αξιοποίησαν στην πράξη τα εθνικά κοινοβούλια αυτά τα δικαιώματά τους, σε τι είδους ζητήματα αξιοποίησαν αυτό το δικαίωμα και πώς λειτουργήσε. Και ε, εγώ έχω αρκετή εμπειρία σε αυτό το τομέα, όχι ενδεχομένω πολύ βαθιά εμπειρία, αλλά στην προηγούμενη βουλευτική θητεία ήμουν αρμόδιο από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματο για τα κοινοβούλια. Οπότε η ιδέα που έχω εγώ και βέβαια θα πρέπει να διαβουλευθώ και με την διευθυντική μα αποστολή είναι η, η, μάλλον η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι δεν λειτουργούν καλά αυτά τα εργαλεία της κίτρινης και πορτοκαλίου κάρτας γιατί υπάρχει ε, αυτή η διαδικασία που προβλέπει μόνο 8 εβδομάδες οπότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε λίγο το κατά πόσο αποτελεί μια ενδεδειγμένη λύση. Επίσης η επικοινωνία μεταξύ των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων είναι δύσκολη οπότε εκείνο που ε, για, υπέρ του οποίου εγώ τάσσομαι είναι μετά από την αξιολόγηση των όσων συμβαίνουν, μετά από την εξέταση των ζητημάτων στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο, αφού εξετάσουμε ε, το κατά πόσο οι αρχές της αναλογικότητας και της επικορικότητας έχουν πράγματι ε, ενσωματωθεί στις αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, αφού λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα εν λόγω εργαλεία. Γιατί είναι θεμελιώδου σημασία στα εν λόγω εργαλεία, έτσι ώστε να ε, χορηγήσουν στα εθνικά κοινοβούλια τις εξουσίες που, τους, τους έχει προσδώσει η συνθήκη της Λισαβόνας και βέβαια μια τέτοια κίνηση θα εκλειφθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια ως μια προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τονώσει, να ενισχύσει τι αρμοδιότητε των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω πως ε, εμείς στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επέτρεπε κάποια ευελιξία στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δηλαδή, ε, συχνά τα Εθνικά Κοινοβούλια ενδιαφέρονται πάρα πολύ ε, για μια τέτοια διακοινοβουλευτική ε, επικοινωνία, αλλά δεν έχουν τα εργαλεία, τα μέσα για να το πράξουν. Οπότε θα μπορούσαμε εμεί από την πλευρά μα να σχεδιάσουμε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούν να αλληλεπιδρούν και μπορούν ακριβώ να αξιοποιούν τι δυνατότητε που έχουν στη διάθεσή του με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο. Νομίζω πω κάτι τέτοιο θα ήταν σημαντικό. Επίση, επιστρέφοντα τώρα ε, στο ζήτημα της ΚΟΣΑΚ, εγώ θα πρέπει να πω πως ε, το εν λόγω φόρουμ της Κοζάκ δηλαδή ε, είναι ε, ένα φόρουμ το οποίο έχει προβλεφθεί για διάλογο μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά έχει μετατραπεί σε ένα είδος ring αγώνων όπου τα εθνικά κοινοβούλια επικρίνουν και μάλιστα κατηγορηματικά και εμφαντικά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο της Κοζάκος το ποιο θα είναι πιο επικριτικό και πιο εμφατικό στις ε, απόψεις του εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πραγματικά δεν θεωρώ ότι το η Κόζακος Φόρουμ αποτελεί ένα ενδεδειγμένο πόνο αυτή τη συζήτηση γιατί τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία έχουν τις, ε, τις ε, λογικές τους τοποθετήσεις, οι οποίες προφανώς μπορούν να είναι επικριτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ε, και μπορούν προφανώς να τις εκφράσουν στο πλαίσιο της ε, ΚΟΖΑΚ. Στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ δημιουργείται ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους όπου το κάθε κοινοβούλιο προσπαθεί ακριβώς να εκφραστεί πιο εμφαντικά σε ό,τι αφορά αυτή την επικριτική στάση. Πράγμα βέβαια το οποίο εν μέρει έχει εξεπαραστεί μέσω των νέων αρμοδιοτήτων που έχουν αποκτήσει τώρα τα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει πάντως να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα και να δούμε ποιε είναι οι μορφέ συνεργασία, επικοινωνία και διαρθρωμένου διαλόγου για να χρησιμοποιήσω έτσι αυτόν τον τόσο διαδεδομένο πλέον όρο του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που τίθενται εδώ και η διατύπωση της γνωμοδότησης θα βασιστεί ακριβώς στα δεδομένα τα οποία εμείς θα διαπιστώσουμε. Ενδεχομένως δηλαδή τώρα να έχω κάποιες εντυπώσεις, κάποιες απόψεις, αλλά όταν θα δω τα στατιστικά στοιχεία, όταν θα δω το τι συμβαίνει στα επιμέρους ελληνικά κοινοβούλια, θα είμαι κι εγώ ε, διατεθειμένος να μεταβάλω τις δικές μου προκαθορισμένες απόψεις. Αλλά υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα ζητήματα τα οποία θεωρώ πως θα πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε δηλαδή ήδη κάποιο κεκτημένο των εισαγωγικών από, την, ε, από τις εκθέσεις Μπροκ και Κασίνη ε, ε, και συμφωνούμε με τις ανησυχίες που εκφράζονται εκεί. και τις εκτιμήσεις δηλαδή που έγιναν στο πλαίσιο αυτών των θέσεων, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιες νέες περιστάσεις, νέες πραγματικότητες τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο πλαίσιο μιας τέτοιας νομοδότησης. Η πρώτη από αυτές, τις νέες παραμέτρους αν θέλετε, είναι πολύ σημαντική για μένα προσωπικά και Ε, τρόπον την να ε, βασίζεται και σε, στην καλή γνώση της ε, πορτογαλικής κατάστασης είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο θεωρώ φρονώ πως αποτελεί ένα από τους κύριους τομείς στους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό δηλαδή που παρατηρώ στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου που λαμβάνει η χώρα και του διαλόγου στο, στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ότι μετά από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν απολέσει την αρμοδιότητά τους σε ό,τι αφορά τα ζητήματα προϋπολογισμού. Αλλά γνωρίζουμε πως ε, τα ζητήματα προϋπολογισμού αποτελούν ε, βασική αρμοδιότητα, βασική εξουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων από το Μεσαίωνα. Ήταν ε, τα, τα επανομαζόμενα κόρτε στην Ιβρική Χερσόνησο, ήταν ε, το, Parliament στην, στο, στην Αγγλία. με άλλες ονομασίες στη Γαλλία και σε, και σε ανατολικές χώρες. Πάντοτε λοιπόν αυτές, αυτά τα κοινοβούλια, οι βουλές είχαν αυτή την αρμοδιότητα της ε, επιβολής ε, φόρων, της αύξησης, η μείωση των φόρων. Πρόκειται λοιπόν για πάρα, ε, μια αρμοδιότητα που βρίσκεται στον πυρήνα, θέλετε, των εξουσιών των Εθνικών Κοινοβουλίων ανέκαθεν. Οπότε, ποιο είναι το δικό μου σκεπτικό ότι θέλω να κάνω σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, να αναφέρω ή να θέσω το γεγονός ότι δεν έχουν προβεί στις δικές τους ενέργειες από την πλευρά, δηλαδή τους, τα εθνικά κοινοβούλια, σε ό,τι αφορά ακριβώς ε, την, ε, την αρμόδια τους, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή παραπονιούνται ότι δεν έχουν απολέσει τη δικιά τους αρμοδιότητα, αλλά δεν έγινε αυτό. Δηλαδή δεν έχουν, θα μπορούσαν να έχουν συμμετάσχει, για παράδειγμα, να έχουν επηρεάσει τον προπολογισμό μέσω της σύνταξης ενός εγγραφού, δεν το κάνουν. Θα συνεχίσουν λοιπόν και έχει ήδη με τη συνθήκη επεκταθεί η αρμοδιότητά τους πολύ περισσότερο από αυτό που ισχυρίζονται. Αλλά αυτό εξαρτάται, δηλαδή η εφαρμογή της αρμοδιότητά τους εξαρτάται από τη διαδικασία έξι του προπολογισμού που ισχύει στο επίπεδο του Εθνικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ε, ενδεχομένω θα πρέπει να προβλέψουν μια μεταβολή του δικού του κανονισμού του, ώστε να υπάρχει ένα είδο, αν θέλετε, εθνικού τριμήνου, το οποίο θα προηγείται του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κάθε φορά. Νομίζω πω αυτό πραγματικά αποτελεί ένα ζήτημα πυρήνα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ένα ακόμα το οποίο έχω συζητήσει και το οποίο, με το οποίο συμφωνεί ο Μπεν Λάγκ που συμμετέχει και στην ε, Επιτροπή και ε, το έχει θέσει σε μια σχετική επιστολή είναι το εξή. Μέσω της ε, συμφωνίας ελεύθερου μπορούμε με τη ΣΥΤΕ έχουμε το ζήτημα που τίθεται σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το κατά πόσο η εν λόγω αυτή η νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα για την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα αποτελεί ε, αντικείμενο μεικτής αρμοδιότητας. δηλαδή, καταρχήν ταξινόμηση των επιμέρων τμήματων αυτής της ε, συμφωνίας και από εκεί και μετά κατανομή αυτών των τμήματων σε εθνική σε ε, ενωσιακή αρμοδιότητα. νομίζω πως θα πρέπει να προβούμε σε μια αξιολόγηση εδώ της κατάστασης γιατί νομίζω πως ελοχεύει ο κίνδυνος να μεταβάλουμε τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τις σχετικές ε, ρήτρε σε κάτι άλλο. Γιατί βέβαια υπήρχαν ρήτρε αυτές που προβλέπουν ε, την στη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω πως θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα στην γνωμοδότηση. Γιατί εάν αρχίσουμε να υιοθετούμε αυτή την άποψη ότι δηλαδή κάθε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου περιλαμβάνει κάποια τμήματα επί των οποίων αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από ψηφοφορία στα Εθνικά Κοινοβούλια, τότε ουσιαστικά θα έχει απολέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εμπορίου. Αυτό είναι ξεκάθαρο κατά τη δική μου άποψη ε, και ε, θεωρώ σημαντικό το γεγονό ότι ο κ. Ζέμπεν Λάγκε θεωρεί και εκείνο σημαντικό το εν ζήτημα και έχει ζητήσει να περιληφθεί στη δική μα εκνομοδότηση. Ούτω ή άλλω, εγώ το είχα ήδη θέσει στο δική μα προσωπικό. Εδώ και στους συναδέλφους ε, υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα νέα ζητήματα που έχουν προκύψει και είναι ε, σχετικά με τη δική μας ε, ε, γνωμοδότηση, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ή συμφωνίες Ελευθερού Εμπορίου, οι οποίες τα οποία ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δική μας γνωμοδότηση. Αρκετά μακρυγόνησε, οπότε θα δώσω την ευκαιρία στους συναδέλφους να με αντικρούσουν και να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Το ΕΛΚ θεωρητικά ήδη μίλησε. Είχα ξεχάσει ότι δεν υπάρχει εδώ σκιώδης του ΕΛΚ. Ο κύριος Κόλμπετ θα πάρει το λόγο, θα κάνω εγώ όμως κάποιες παρατηρήσεις. Η κυρία Περές που είναι σκιώδης εισηγητριά μας για το θέμα αυτό δεν είναι παρούσα. Θα έχει τη δυνατότητα να σας παρουσιάσει τις παρατηρήσεις της όμως. Μόλις έχουμε συγκεκριμένο κείμενο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ραντζέλ, διότι νομίζω ότι αναλύσατε τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προκύπτει σαφώς από την εξέλιξη των ε, θεσμικών συστημάτων ότι υπάρχει μια αποδυνάμωση των κοινοβουλίων σε σχέση με τις κυβερνήσεις και αυτό παντού. Οπότε αυτό έχει συνέπειες όσον αφορά τις δικές μας σχέσεις με αυτά τα εθνικά κοινοβουλία. Έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε αμυντική στάση, είναι στριμωγμένα όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους μέσα στην ίδια τους τη χώρα αμυντική στάση. Πάνω σε αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, στο κείμενό μας ασχολούμεθα με τα όσα είναι ισχύοντα δυνάμει των συνθήκων. Και επίσης Βλέπουμε και τι προοπτική ξανήγεται, φύγεται και αυτό. Θα δούμε τι σενάρια ξενεύονται για το μέλλον, τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, πώς μπορεί ακριβώς αυτές οι σχέσεις με την Κοινοβούλια να βελτιωθούν. Όπως ξέρετε, έχω διατελέσει πρώτα στην Επιτροπή των ε, περιφερειών, είναι και τα θέματα της ε, επικουρικότητας, είχε γίνει, υπάρχει και νομολογία τέλος πάντων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο το να μπορέσει κανείς να περάσει κάποια νομοθετική πρόταση εάν αυτή ε, έρχεται σε σύγκρουση με την επικουρικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν τις προτάσεις, αξιολογώντας, ζυγίζοντας το τι ισχύει. και πάντα διαμορφώνει τις προτάσεις ακριβώς άπαξ και δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση με τα ισχύοντα στις συνθήκες και δυνάμει αυτών. Επομένως αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, η συγκυρία, οι δυσκολίε που υπάρχουν και να δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα. ο πλευράς, εμείς εδώ είμαστε ένα νομοθετικό σώμα. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς κανείς μπορεί να επιτεθεί ε, και να πλήξει την επικουρικότητα και άρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι και τόσο μεγάλα τα περιθώρια προς τούτο. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι δυνατότητες δίνονται από το ίδιο το σώμα του κειμένου, ας πούμε, των συνθήκων. Και έτσι να δει κανείς τι γίνεται από πλευράς ε, αξιολόγησης όσον αφορά την ουσία των προτάσεων. Αυτό έχει ζητηθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό αφορά η προβληματική και η πολεμική η πράσινη κάρτα δηλαδή. Υπάρχει πρόθεση συνεργασίας και άρα βρισκόμαστε ενώπιον του παραδόξου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδομηθεί από τα βασικά θεσμικά όργανα όπου συμμετέχουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, έχουμε επίσης δύο επιτροπές που εκπροσωπούν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά επίσης ε, και ε, κάποια, την κοινωνία, διάφορους κλάδους της οικονομίας. Έτσι γίνεται η εκπροσώπηση. Άρα αυτό να σκεφτούμε όσον αφορά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής θεσμικής αρχιτεκτονικής. Να δούμε τι γίνεται. Τις επικαλύψεις που τυχόν έχουμε σήμερα στο Συμβούλιο, εκεί που ε, έχουμε διπλή εκπροσώπηση ούτως επί των κρατών μελών. Έτσι να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Να δούμε τι αρμοδιότητες προβλέπουν για τα κράτη-μέλη που είναι διάφορες, πολλές. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Κόρμπετ. Ε, για ποιο τους κυβέρνηση στη θέση του Συμβουλίου, λέει στον κύριο Κόρμπετ ο ομιλήτρια. να δούμε μόνο τι δεν πάει καλά, τι δεν δουλεύει καλά. Αυτό είναι το καθήκον μας, αυτό πρέπει να κάνουμε με αυτή την έκθεση. Άρα είναι σωστό το πώς λειτουργούν οι διακοινοβευτικές ε, αντιπροσωπείες και επιτροπές αλλά θα πρέπει να δουλέψουν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτόν τη λειτουργία να ε, εξετάσουμε, όχι ότι τα πάνε άσχημα, αυτές οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές. Ασχολούνται και με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα είναι χρήσιμη μια τέτοια ιδέα. αυτές, οι, αυτές οι ημερίδες 13 Φεβρουαρίου, ξέρω εγώ τι άλλο λέμε, να δούμε πώς θα αποδώσουν περισσότερο αυτή η προβληματική για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, για τις οικονομικές πολιτικές, γενικά ε, τα χρηματοοικονομικά της Ένωσης. Νομίζω ότι έτσι μπορεί να διορθωθεί καλύτερα η σχέση Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Επομένως έτσι να δούμε πώς θα έχουν ένα πιο άρτιο νομοθετικό οπλοστάσιο του Εθνικά Κοινοβούλια. Και επομένως να μην έχουμε μόνο ε, κουβέντες και συζητήσεις να έχουμε τις πράξεις των Εθνικών Κοινοβουλίων μέσα ε, ε, από τα οποία, από τις πράξεις να εκφράζεται η γνώμη τους, η άποψή τους, η θέση τους. Έτσι να προβάλλονται αυτές οι ξεκάθαρες, κρυστάλλινες ε, θέσεις και τοποθετήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό θα είναι χρήσιμο. Επίσης, ίσως θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα ισχύοντα τώρα ε, νομοθετικά μέσα και εργαλεία. αυτές οι 8 εβδομάδες πως που γίνεται να παραταθούν, να γίνει μεγαλύτερη η περίοδος. Πολλά εθνικά κοινοβούλια αποτελούν μια πλειοψηφία σε σχέση με το ότι θέλουν να υπάρξει αναθεώρηση, να υπάρξει αξιολόγηση του θεσμικού πλαίσιου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα και φυσικά και η ίδια μας η Επιτροπή. Θα πρέπει να δούμε διακοινοβουλευτικά, δηλαδή σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις ε, προτάσεις της εκθεσής σας και να συνεξετάσουμε τα εθνικά κοινοβούλια για το πώς μπορεί καλύτερα να οργανώσουμε και να διαρθρώσουμε αυτά τα οποία δυνάμει των ισχυουσών συνθήκων ισχύουν ούτως υπήν. Έτσι επομένως να τα σκεφτούμε, να προβληματιστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια και έτσι να καταλήξουμε σε καλύτερες σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια με την αλλαγή του πλαισίου. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό. Πώς θα δημιουργηθούν οι μέλουσες σχέσεις με εκείνα τα κοινοβούλια. Έχουμε και το κείμενο Φερχόφστατ, έτσι και αλλιώς. Αλλαγή των λοιπόν των θεσμικών εργαλείων και βελτίωση των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Ραντζέλ για την εισαγωγή που μας κάνατε. και για την άποψη ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις ε, προτού αποφασίσουμε τι μορφή θα πάρει η έκθεση. Ο κύριος Ράντζελ ανέφερε την θεσμική ζήλια ανάμεσα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να ξεπεραστεί και ίσως το κλειδί για να επιλύσουμε την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τα ε, κοινοβούλια των κρατών μελών. Είναι ε, επικίνδυνη η υπερβολική αποκέντρωση, όπως είπε ο κύριος Βαντζέλα, αλλά και η υπερβολική συγκέντρωση είναι εξίσου επικίνδυνη. Ελπίζω κάθε μεταρρύθμιση να οδηγήσει σε περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη μία και των Εθνικών Κοινοβουλίων από την άλλη. Δύο τομείς θα πρέπει να αναφέρουμε. Που επίσης ανέφερε ο κύριος Ραντζέλ. Μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων. Διότι φυσικά τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους από μόνα τους, αλλά υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, έγινε συνάντηση των κοινοβουλίων των χωρών D4. Αλλά καλό θα είναι να υπάρξει μια πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο. Επίσης, να εφαρμόσουμε σωστά τις διαδικασίες της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τίποτα δεν υπονομεύει περισσότερο την εμπιστοσύνη από προγράμματα που δεν πραγματοποιούνται. Κάτι τέτοιο βλάπτει την αξιοπιστία των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και τι γίνεται όσον αφορά τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Ε, βάσιμες ε, παρεμβάσεις των, των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν λαμβάνονται υπόψη. Έχουμε λάβει διάφορες ε, προσφυγές από τα Εθνικά Κοινοβούλια χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην οδηγία. Τα εργαλεία λοιπόν που έχουν δοθεί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε επίσης να τονίσει περισσότερο την αρχή της επικουρικότητας στις εργασίες του. Μία από τις τροπολογίες ε, για την έκθεση του κυρίου Κόρπετ προωθεί τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου στον τομέα της επικουρικότητας. Μέχρι τώρα είχαμε αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Γιούρη. Θα μπορούν όμως και οι πολιτικές ομάδες ε, να εφαρμόζουν την ε, αρχή αυτή στις εργασίες τους. Ε, και τίθεται και το θέμα της επικοινωνίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρότεινα να ακολουθήσουμε την οδό της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα, Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν. Ελπίζω να μπορέσουμε να οργανώσουμε δημόσια ακρόαση με συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ίσως να μπορούσαμε να οργανώσουμε και κάποιες διασκέψεις, κάτι τέτοιο θα μας ε, επέτρεπε να δώσουμε την ε, τελική μορφή στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ από την άλλη. Δεν υπάρχει κανείς από την ΚΟΕ. Παρακαλώ, ο Χέρμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την έναρξη μιας συζήτησης η οποία νομίζω ε, θα μας απασχολήσει επί εβδομάδες ε, ή και μήνες, διότι είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Αναρωτιέμαι γιατί ήδη έχουμε μια τέτοια εισβάθος συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι με φόντο τις ε, πολύπλοκες ε, οικονομικές καταστάσεις. Πρώτη φορά συνειδητοποιούμε τώρα ποιος αποφασίζει και σε τι επίπεδο σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική. Και οι πολίτες ε, νιώθουν ανασφάλεια, διότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και τώρα με τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, συμφωνήσει πάνω στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο είναι μάλλον εφελώδες και έτσι ως Κοινοβούλιο έχουμε αντιμετωπίζουμε διτή πρόκληση. Από τη μία θα πρέπει να σκεφτούμε και συμφωνώ με ε, τον προλαλήσαντα, πρέπει να έχουμε ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια και όλους ε, τους άλλους ε, ενδιαφερόμενους σε εθνικό επίπεδο και από την άλλη θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε με τις απόψεις αυτές τις δικές μας διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όπως είπε και η συνάδελφος Μπρέσο, θα πρέπει να δούμε ότι χρειαζόμαστε μηχανισμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας περισσότερο από αυτούς που έχουμε μέχρι τώρα. Και έτσι περνώ στην τρίτη μου παρατήρηση. Δεν είναι ακριβώς ε, υποχρέωση των ε, κυβερνήσεων να δώσουν το ρόλο που πρέπει στα εθνικά κοινοβούλια, στα ευρωπαϊκά θέματα. Όταν ε, συνέρχονται οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπουργοί, αντιπροσωπεύουν την θέση των κυβερνήσεων. Αλλά η θέση αυτή πώς έχει διαμορφωθεί. οι κυβερνήσεις συχνά δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη θέση των ε, εθνικών κοινοβουλίων σε εθνικό επίπεδο και έτσι δημιουργούνται και ένα το θέμα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί ο εισηγητής θίγει το ερώτημα πόσο δημοκρατικό και σε πόσο δημοκρατικά διαμορφώνονται τελικά οι θέσει μας. Και συμμετέχουν οι πολίτες ε, στην διαμόρφωση της νομοθεσίας, ε, διότι για νομοθεσία πρόκειται. Για παράδειγμα, οι εμπορικές ε, συμφωνίες που συνάπτονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρακτικές συνέπειες στα κράτη-μέλη και βρίσκω ενδιαφέρον το να έχουμε μία συζήτηση σχετικά με την ε, εφαρμογή των ε, άρθρων της συνθήκης της Λισαβόνας ε, με τις οποίες εκχωρείται η κυριαρχία των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η σχέση μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και του εθνικού ενδιαφέρον. Είναι αυτό που ε, συνέβη και έχω εγώ 25-26 ερωτήσεις σε, σε τι βαθμό λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πόσο λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές θέσεις ε, ακόμα και σε το μίσο που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι αντιδράσει στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ περισσότερη ανταλλαγή ε, πληροφοριών και απόψεων ε, με τα εθνικά κοινοβούλια. Χρειαζόμαστε περισσότερη προετοιμασία κατά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων. Και εγώ και η Ισκιώδης, ε, ε, η συγγήτριά μας η Μπάρβαρα Σπινέλη, προσβλέπουμε με πολύ ενδιαφέρον ε, τη συνέχιση των εργασιών. Ευχαριστώ, Μαξ Άντερσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα για τη δημοκρατία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τις τελευταίες μέρες είναι η τεράστια μεταφορά εξουσιών ε, από εθνικά κοινοβούλια στις κυβερνήσεις. Διότι οι θέσεις των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαμορφώνονται πια εντός των κοινοβουλίων. Οι κυβερνήσεις συμμετέχουν ε, στις ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου και μπορούν να επηρεάσουν ε, την κατάσταση, αλλά δεν χρειάζεται να ακούνε τι λένε τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι στο Συμβούλιο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μία από τις συνέπειες της, των τελευταίων τροποποίησεων της συνθήκης ήταν ακριβώς η μεταφορά εξουσίας ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να οικοδομήσει νέα κοινοβουλευτική εξουσία που να συγκρατεί το Συμβούλιο και έχει γίνει αυτό σε κάποιο βαθμό. Τα Εθνικά Κοινοβούλια όμως έχασαν από όλη αυτή τη διαδικασία. Οι κυβερνήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν συνεργάζονται τόσο πολύ μεταξύ τους. Πώς μπορούμε λοιπόν ε, να επαναφέρουμε την ισορροπία στην κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι οι προτάσεις ε, που υιοθετήθηκαν στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, σχετικά με την κίτρινη κάρτα, τον έλεγχο της επικουρικότητας κλπ. αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά πρώτον δεν λειτουργούν πολύ καλά ακόμα και χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. Τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια ούτε καν κάνουν τον κόπο να πάρουν στα σοβαρά τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Μερικά κοινοβούλια το κάνουν αυτό, αλλά για να λειτουργήσει η διαδικασία αυτή, για να του λειτουργήσει τόσο καλά ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να να δαπανίσουν το, το δυναμικό που χρειάζεται, θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Εάν λοιπόν ασχοληθούμε εμείς, ε, ίσως ασχοληθούν και τα εθνικά κοινοβούλια. Τώρα που τα εθνικά κοινοβούλια δεν παίρνουν πολύ στα σοβαρά αυτή τη ε, διαδικασία, ε, δεν υπάρχει και κίνητρο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δίνουμε τις προσπάθειές μας. Κάναμε προσπάθειες αλλά δεν αρκούσαν. Μάλλον χρειαζόμαστε πιο χαμηλό κατόφλι για την χρήση της κίτρινης κάρτας ε, για να κίνητρα στα εθνικά κοινοβούλια τη χρησιμοποιούν και θα πρέπει να βελτιώσουμε και την επικοινωνία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων. Επίσης, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν πολύ πιο νωρίς στην πολιτική διαδικασία. Γι' αυτό Υπάρχει πρόταση της κίτρινης κάρτας, υπάρχει όμως ε, και η πρόταση της πράσινης κάρτας, ώστε να μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Επίσης, όσον αφορά την αμοιβαία εμπιστοσύνη, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και από τη μία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άλλη και μάλιστα αμοιβαία ε, έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να επαναφέρουμε την ισορροπία ανάμεσα στις κυβερνήσεις ε, και τα κοινοβούλια. Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια θα πρέπει να συνεργαστούν για να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Περβάνω Περές. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όμως και τον φίλο κύριο Ραντζέλ, τον εισηγητή μας. Ε, που δεν ήμουν πιο νωρί γιατί είχα κάποια άλλη υποχρέωση και με μεγάλη προσοχή μελέτησα όσα προτείνει στο κείμενό του ο εισηγητής και θα ήθελα χρησιμοποιώντας ό,τι πιστεύω για το θέμα ότι μπορώ να συμβαλώ ως εξή. λέμε και τονίζουμε ότι το άρθρο 3 αποτελεί πρόοδο σε σχέση με άλλες μορφές συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όμως, τελικά, αυτό το οποίο λείπει είναι η διευκρίνηση, το ξεκαθάρισμα του ρόλου όλων των πλευρών όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Τα ξέρουμε αυτά, έχουμε επεξεργαστεί μαζί το κείμενο που αφορούσε τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Άρα προσοχή στη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια να μην χάσουμε το εγκάρσιο, την ουσία που είναι ο δημοκρατικός έλεγχος. Αυτός επιτελείται καλύτερα όταν ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Όταν ο καθένας λαμβάνει την απόφαση που οφείλει να λάβει στο επίπεδό του. Αυτό είναι το σημείο συνάντησης των μεν με τους δε. Πολύ σημαντικό βέβαια να υπάρχει αυτή η εμπλοκή, αυτό το δίκτυο, η δικτύωση δηλαδή. Αλλά προσοχή μην φτιάχνουμε κάποιες δομές που οδηγούν στη σύγχυση. Γιατί σύγχυση και μόνο θα βασιλεύσει αν δεν μπορεί να ασκήσει κάποιος κοινοβουλευτικός τα καθήκοντά του. Όταν λοιπόν στο πλαίσιο ευρωπαϊκή οικοδόμηση καθορίζουμε ποιο είναι ο ρόλο του Εθνικού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να βρούμε πότε θα πρέπει να δράσουν αυτό το κοινοβούλια. Επομένω, αυτό είναι το βασικό όπλο που έχουν σήμερα. Είναι ένα, ε, ένα εργαλείο αρνητικό ούτω ή Αυτό, η υπόθεση αυτή τη κάρτα, τη πράσινη κάρτα κλπ. Να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Καλά, αυτό θα μπορούσε να αφορά και αναθεώρηση των ίδιων των συνθηκών. Άρα, για μένα αυτό είναι ο μπούσουλα. Το πώ θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τι κάνει, τι, δουλειέ, τι αρμοδιότητε οφείλει να κάνει η κάθε πλευρά. Τώρα για τα οικονομικά και, και τα λοιπά, αυτά τα ξέρει ο εισηγητή πρόεδρο. Θα πρέπει να φύγει ο Παλαιός να τον πρόεδρο Σούλσκ. Καλά, θα το, σημειώσουμε και θα το διαβιβάσουμε. Αλλά τέλος πάντων το θέμα θα ζητηθεί μέχρι το Μάιο του 2017. Θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Ραντζελ. Συμπαθάτε με αλλά έχει τη διάσκεψη των Προέδρων. Σε 10 λεπτά ο Πρόεδρος. Και μου είπε στις παρατέταρτο να πάω να τον συναντήσω. Απλώς να σας πω ότι Όλα αυτά που άκουσα είναι πολύ σημαντικά. Καλή ιδέα αυτή η πράσινη κάρτα για την οποία όλοι μίλησαν. Και άλλο σημαντικό είναι ο διάλογος με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Για συγκεκριμένα θέματα μεταξύ των οποίων είναι και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. πολύ πιο αποτελεσματική είναι μια τέτοια συνεργασία παρά η συνεργασία που γίνεται τώρα στην Κόζακ. Οπότε, νομίζω δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τι μοντέλο θα παρεμβαίνουμε στο συνταγματικό πλαίσιο που διέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η κατοβουλία εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Δηλαδή το το συμβουλευτό είναι το μοντέλο το οποίο επιβλήθηκε και δύναμη του Αμερικανικού Συντάγματος επί Ρούσβελτ. Οπότε, στη Γερουσία έχουμε βουλευτές και στις, ε, στην Κατοβουλή Βουλή έχουμε τους εκπροσώπους, τους εθνικούς αντιπροσώπους τέλος πάντων κάτω έχουμε και τι εκλογέ, να δούμε τι θα γίνει. Επίση στην Ελβετία ε, οι άνθρωποι εκλεγούν του ε, αντιπροσώπου του. Ε, από τα μέλη των κοινοβουλίων του κάθε κρατηδίου της κάθε περιοχής. Να, σας παραπέμπω στο κείμενο Φερχόφστατ. Άρα, θα πρέπει να γυρθούμε στα πλαίσια του ισχύοντος συνταγματικού πλαίσιου. Τέλος πάντων, συγγνώμη, θα φύγω, αλλά θα είμαι να τα συζητήσουμε άλλη φορά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει τώρα να φύγω. We Thank you very much. I understand why you have to Σας ευχαριστούμε και ε, αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να φύγεις αλλά θα χάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, πάντως Μπορεί να τη δεις μέσω web streaming την υπόλοιπη συζήτηση. Θα σε βάλω και εγώ στο να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον συνάδελφο για τη δουλειά που ήδη έχει κάνει. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα τη θεσμική ζήλια που αναφέρθηκε, δεν ξέρω αν πρόκειται για τον πλέον εύστοχο. Ουσιαστικά ε, ε, υπενήσεται κάτι αυτό ο όρο. Ε, συμφωνώ καταρχήν στο αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος ότι δηλαδή η ΚΟΖΑΚ μπορεί να αποτελέσει ένα φόρουμ όπου υπάρχουν τριβές αλλά αυτή είναι και μια ε, εντελώς φυσιολογική σχέση μεταξύ διαφορετικών κέντρων εξουσίας αν θέλετε. Δηλαδή όταν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσία που αλληλεπιδρούν τότε θα υπάρξουν κάποιες συγκρούσεις. Ε, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό αυτό. Μπορούμε να το ονομάσουμε αν θέλετε θεσμική ζηλιά αλλά το θεωρώ πως κάτι το φυσιολογικό. Αν υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση τέτοια εξουσία τότε θα πρέπει να προβλέψουμε ε, έναν τρόπο επίλυσης αυτών των διαφόρων και συγκρουσιών. Και τίθεται το ερώτημα του πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την επίλυση. Ε, για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε πολύ πιο ε, σοβαρά το τι κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπότε θέτω σε εσά ένα ερώτημα. Θα μπορούσαμε να οθετήσουμε μια πρακτική πρόσκληση των Εθνικών Κοινοβούλιο για να συμμετάσχουν στη σχετική συζήτηση. Δεν ξέρω αν είχατε ήδη προσκαλέσει τα Εθνικά Κοινοβούλια στο να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση, αλλά δεν βλέπουμε πολλούς εκπροσώπους, οπότε δεν ξέρω, ίσως υπάρχει ένα ζήτημα επικοινωνίας, αναποτελεσματικής. Εγώ βέβαια δεν ήμουν ποτέ μέλος ε, του Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά υπήρξα, είχαμε επαφή και νομίζω πως ε, η εντύπωση που έχω είναι ότι η, Επιτρο... η, Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή δηλαδή και για ε, ευρωπαϊκά ζητήματα είναι ε, πολύ ενδιαφέρουσα ε, αλλά δεν βλέπουμε να παρακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τα όσα συμβαίνουν εδώ στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από εκεί και μετά θα ήθελα να αναφέρω ότι η αυξανόμενη δυσαρέσκεια από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων αποτελεί ένα πρόβλημα τόσο για εκείνα όσο και για μας. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αίσθηση σε εθνικό επίπεδο, και να το πω όμα, ότι το, εθνικό, το Ευρωπαϊκό Συνόμιο Κοινοβούλιο έβαλε υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας. Και ε, μετανιώνουν ότι δεν παρενέβησαν εγκαίρως και αυτή είναι η αίσθηση την οποία εγώ αποκομίσω από διάφορες απαντήσεις σε ε, που δόθηκαν όταν δηλαδή ε, δημοσιεύτηκε πλέον η συνθήκη της Λισαβόνας ε, και νομίζω πως είναι πολύ σωστό αυτό που ανέφερε ο Πάολο δηλαδή ότι υπάρχει ένα άλλος ανταγωνισμού μεταξύ των Αθηνικών Κοινοβουλίων ως προς το ποιος μπορεί να είναι ο δημήτρης κριτικός μας. Τώρα, νομίζω πως στην πλήρη του προβλήματος βρίσκεται ότι δεν έχουμε απλώς διαφορετικά κέντρα αν θέλετε εξουσίας, αλλά έχουμε και διαφορετικούς βαθμούς νομιμοποίησης αυτών των κέντρων εξουσίας. Και το ζήτημα που συζητήθηκε επανειλημμένα στο πλαίσιο της δικής μας επιτροπής, για παράδειγμα και στο πλαίσιο της συζήτησης έκθεσης Κασίνη στο κοινοβούλιο της προηγούμενης ε, θητείας, είναι το ε, ε, κατά πόσο πράγματι μειώσαμε την νομιμοποίηση των Εθνικών Κοινοβουλίων προκειμένου να αυξήσουμε τη δική μας νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, γιατί φαίνεται να το έχουν αντιληφθεί αυτό σε κάθε περίπτωση στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ένα ακόμα σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτήν την ε, μετακίνηση αν θέλετε, της που ανέφερε ο κύριος Άντερσον ε, ναι, υπάρχει μια γενικότερη αναδιανομή, αν θέλετε, ανακατανομή των εξουσιών, ε, η οποία λαμβάνει η χώρα κατά τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δηλαδή, κατευθύνεται από τους νομοθέτες προς τους ε, κοινωνικούς φορείς, αν θέλετε, δηλαδή και στου στους κοινωνικούς εταίρους, οργανώσει οργανώσεις και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, οι νομοθέτες είναι λιγότερο σημαντικοί από ό,τι ήταν κάποτε πριν από 50-60 χρόνια, πράγμα το οποίο τους δυσαρεστεί. Ε, και κάτι ακόμα που ανέφερε ο συνάδελφος ό,τι αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ε, αντιλαμβάνομαι το πώς η ε, πορτοκαλί κάρτα η, η, η, τρίτη φορά όπου ουσιαστικά δόθηκε η κίτρινη κάρτα και αγνοήθηκε παντελώ, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερη δυσαρέστια και τελικά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το να υπάρξει κόκκινη κάρτα. Ε, και νομίζω πως αυτό είναι σημαντικό δηλαδή και απόψη διακυβέρνησης ε, ε, είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά και 11 κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω πως σε σχέση με αυτό το ζήτημα μπορούμε να αντιληφθούμε πώς θα σκεφτούν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν μας παίρνει στα σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο κατηγορηματικοί ούτως ώστε να μας πάνω στα σοβαρά. Ναι. Ε, θα πρέπει όμως να θυμηθείς ε, ότι υπήρχαν εκπρόσωποι στο πλαίσιο της συζήτηση ε, για την συνθήκη και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μάλιστα και από τις δύο βουλές όπου υπήρχαν. Οπότε συμμετείχαν στη διαδικασία διατύπωσης αυτής της συνθήκης. Ο λόγος του Ρίτσαρτ Κόμπ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε για την ζήλια ανάμεσα στα κοινοβούλια και αν υπάρχει κάτι τέτοιο νομίζω ότι αυτό συμβαίνει εν μέρη επειδή ε, το Κοινοβούλιο τροποποιεί και ε, κατά καιρού απορρίπτει την νομοθεσία που υποβάλλεται σε αυτό, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια δεν το κάνουν αυτό. Ε, εάν, για παράδειγμα, την Βουλή των Κοινοτήτων, συχνά έχουν πολύ έντονες συζητήσεις, πιο έντονες από τις δικές μας, αλλά πολύ σπάνια τροποποιούν νομοθεσία που έχει υποβάλει η κυβέρνηση. Ε, αν θυμάμαι καλά, μία φορά έγινε αυτό στην ε, τελευταία θητεία. Ε, τρόμος, φόβος και τρόμος που υιοθετήθηκε μία ε, τροπολογία που δεν άρεσε στην κυβέρνηση. Έχουμε την εκτελεστική εξουσία, έχουμε την πλειοψηφία που ε, ψηφίζει αυτά που προτείνει η κυβέρνηση δημοκρατικά όλα αυτά, αλλά εδώ στο Κοινοβούλιο σπάνιο λαμβάνουμε ένα σχέδιο πρότασης ε, που να μην το τροποποιήσουμε. Ίσως λοιπόν ε, αυτό να οδηγεί σε κάποια ζήλια όσον αφορά τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας και της πορτοκαλί κάρτας. Αυτό υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Νομίζω ότι θα έχουν υιοθετηθεί ίσως και χίλια νομοθετήματα στο διάστημα αυτό. Ούτε μία φορά δεν φτάσαμε το κατόφλι για την κίτρινη κάρτα. Τρεις περιπτώσεις ε, είχαμε κίτρινης ε, κάρτας για απόρριψη πρότασης για την ε, λόγω επικουρικότητας. Ε, τρεις φορές ε, έχει επιτευχθεί μειοψηφία, όχι πλειοψηφία όπως στην περίπτωση της πορτοκαλί κάρτας. Τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια τώρα έχουν το σύστημα IPEC για να συνομιλούν μεταξύ τους, για να ενημερώνουν το ένα το άλλο, το τι κάνει. Οχτώ εβδομάδες δεν πια και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στι ε, περισσότερε περιπτώσει νομοθετικών προτάσεων η επικουρικότητα φαίνεται να μην είναι πρόβλημα. Η η... το... το περιεχόμενο μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, όχι όμω η επικουρικότητα. Και σκεφτείτε, το λογικό είναι. Για να υιοθετήσει κανεί οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται πέρα από την έγκριση του Κοινοβουλίου και την έγκριση του Συμβουλίου, όπου συμμετέχουν εθνικοί υπουργοί που λογοδοτούν στα εθνικά κοινοβούλια εθνικοί υπουργοί που δεν θα επιλέξουν απαραίτητα την νομοθεσία σε, εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν αρκεί η νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Και δεν χρειάζεται απλά πλειοψηφία, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Θα πρέπει δηλαδή η ειδική πλειοψηφία των Υπουργών να συμφωνεί ότι ναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα που εμποδίζει την υπερβολική συγκέντρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη, όσο προχωράει ο χρόνος, όλο και περισσότερες νομοθετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν να κάνουν με την τροποποίηση ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, και δεν αποτελούν νέα νομοθεσία σε νέο τομέα. Έτσι λοιπόν η συζήτηση για το αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη γίνει εδώ και πολλά χρόνια και τώρα απλά τροποποιούμε, επικαιροποιούμε, με προσαρμόζουμε ε, στις ε, νέες συνθήκες. Ε, ακόμα και αυτό βέβαια μπορεί να γύρει θέματα επικουρικότητας, αλλά όχι τόσο συχνά. Για τους δύο αυτούς λοιπόν λόγους ε, δεν νομίζω ότι ο μηχανισμός για την επικουρικότητα με την κίτρινη κάρτα και την πορτοκαλή κάρτα ε, θα κινητοποιούνται συχνά. Είναι σημαντικό διασφαλιστικό μέτρο, ε, έχει καλώς. Πιο σημαντικό είναι στη προθεσμία 8 εβδομάδων που δίδεται στα Εθνικά Κοινοβούλια, τα κοινοβούλια να διαμορφώσουν στο διάστημα αυτό την, ε, την άποψη του Υπουργού τους στο Συμβούλιο και όχι απλά να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τις θέσεις των Υπουργών τους στις Βρυξέλλες. Κάποια κοινοβούλια, από ό,τι γνωρίζω, το κάνουν αυτό καλύτερα από άλλα. Ο κύριο Άντεσον να με διορθώσει αν κάνω λάθο. αλλά νομίζω ότι στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φιλανδία κάθε υπουργό ε, που και Γερμανία ακούω και στι χώρε τη Βαλτική. Όποιο υπουργό ε, έχει να πάει την άλλη εβδομάδα στι Βρυξέλλε, σε τούτη την εβδομάδα θα επισκεφτεί την σχετική επιτροπή του Κοινοβουλίου και θα λέει ότι αυτό το θέμα έχουμε στη μέση διάταξη, αυτή είναι η θέση που σκοπεύω να ε, κρατήσω και δίδεται η σχετική εντολή. Έτσι λοιπόν ε, λαμβάνουν παρατηρήσει επί τη ουσία, ε, διότι η επικουρικότητα σπάνια είναι πρόβλημα. Αλλά εθνικά κοινοβούλια δεν κάνουν τίποτα τέτοιο. Τίποτα δεν του σταματάει από το να το κάνουν. Ε, είναι θέμα εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών. Δεν μπορούμε λοιπόν να του επιβάλλουμε κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να του πούμε πώ θα οργανώσουν τι εργασίε του. Κάποια εθνικά κοινοβούλια λοιπόν που ανησυχούν για το θέμα αυτό, μήπως θα πρέπει να επανεξετάσουν τις δικές τους διαδικασίες. Όσον αφορά τις ε, κοινοβουλευτικές ε, διασκέψεις, σύμφωνο με αυτούς ε, που λένε ότι το άρθρο 1 και το άρθρο 13 του Συμβόλου Σταθερότητας λειτουργούν καλύτερα, αλλά οι συνέπειες αυτές ε, πιο μεγάλη σημασία έχουν ε, ως ευκαιρίες δικτύωσης ε, παρά ως διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δεν δίνεται η αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων Ε, το θέμα είναι λοιπόν ε, τα εθνικά κοινοβούλια πώς δίνουν εντολή στους υπουργούς, τους, που ε, τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτούς τους φορείς. Δίνουν εντολή στους υπουργούς τους, αλλά δεν μπορούν να δώσουν και εντολή σε μια ομάδα βουλευτών που θα πάει σε έναν από αυτούς τους φορείς. Αποτελούν όμως αυτά ευκαιρίες για δικτύωση, για επαφές σχεδόν τελευταία παρατήρηση, συμφωνώ με τον κύριο Ραντζέλ. ότι έτσι όπως εξελίσσεται το εμπόριο κινδυνεύουμε να αφαιρέσουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο την αρμοδιότητα και να την επαναφέρουμε στο εθνικό επίπεδο ακόμα και η Συμφωνία ΣΥΤΑ απαιτεί ε, έγκριση από 40 διαφορετικά κοινοβούλια, τα 7 από αυτά βρίσκονται στο Βέλγιο οι φορείς τέλος πάντων. Και έτσι μπορούμε να φτάσουμε στην γελία κατάσταση. Ε, το Κοινοβούλιο της, Γερμανικής, ε, της Γερμανόφωνης Μειονότητας ε, στο Βέλγιο που εκπροσωπεί 30.000 ανθρώπους να μπλοκάρει το σύνολο της συμφωνίας που αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Και τελευταία μου παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Κοινοβούλιο διεξάγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα δικαστική υπόθεση κατά του Κοινοβουλίου, διότι το Κοινοβούλιο ε, ε, σκοπεύει ε, να κινητοποιήσει τη διαδικασία του άρθρου 50 για το Brexit χωρίς ψηφοφορία στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αποκλειστικά δηλαδή με βάση το αποτέλεσμα του συμβουλευτικού δημοψηφίσματος που έγινε πριν μερικούς μήνες. Η επίκληση του άρθρου 50 μπορεί μέσα σε δύο χρόνια να οδηγήσει σε έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι που επηρεάζει και τους ε, πολίτες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου λοιπόν έχουμε αυτή την προσφυγή επειδή δεν υπήρξε κοινοβουλευτική εντολή. Όλοι θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ρίτσαρντ. όσον αφορά τις δραστηριότητε των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, σχετικά με τα σχέδια νομοθεσίας ε, των κυβερνήσεών τους. Ε, νομίζω ότι αυτό διαφέρει στην Ευρώπη. Η Σιλβί Κάουφμαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι τα όσα είπε μόλις τώρα ο Ρίτσαρντ ε, γιατί με κάλυψε στα σχόλια που ήθελα να κάνω. Κατά συνέπεια ε, δεν θα με ε, Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αρχής της επικουρικότητας, η Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο μία έκθεση και εμεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου την αξιολογούμε σε ό,τι αφορά δηλαδή την εφαρμογή ακριβώ αυτής της αρχής. Ίσως ε, λοιπόν οι συγκητές μας ε, θα έπρεπε να ε, εξετάσουν αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με αυτή την εφαρμογή. Εκείνο πάντως που με εκπλήσει κάθε φορά στο πλαίσιο του διαλόγου που γίνεται για την βολή της αρχής της επικορυγότητας πόσο διαφορετικά αξιολογείται η πρόταση της Επιτροπής από τα διαφορετικά εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή ένα κοινοβούλιο μπορεί για παράδειγμα να δείξει μια κάρτα και ένα άλλο όχι. Και νομίζω πως ο συνάδελφος ε, ε, το απάντησε πολύ σωστά αυτό το ερώτημα. Υπάρχει διαφορετική πολιτική αξιολόγηση ε, της, της αρχής της επικουρικότητας. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα και διαφορετικές δηλαδή πολιτικές συγκυρίες στα επιμέρους εθνικά κοινοβουλία και από αυτό εξαρτάται και η απόφαση που λαμβάνουν σε ό,τι αφορά ε, και η αξιολόγησή του σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση της αρχής της Ε, Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά τη χάραξη τη ευρωπαϊκή ε, πολιτική. Νομίζω πω ο συνάδελφο Σόλτ έθιξε εδώ κάτι πολύ σημαντικό και θεωρώ πως θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αυτό της έκθεσης, δηλαδή το πόσο ευρύ είναι το πεδίο ε, και το, πόσο μεγαλώνει τον εύρο των δικαιωμάτων που έχουν ε, αποκτήσει τα εθνικά ε, κοινοβούλια για την ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή μία συμφωνία η οποία ε, συνάφθη ε, μεταξύ της Κάτω Βουλής και της ε, Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας στο πλαίσιο κύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία ακριβώς εγγυάται τα δικαιώματα της Κάτω Βουλής ως προς το, τα όσα συμβαίνουν εδώ, στο επίπεδο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα δικαίωμα λοιπόν το οποίο έχει θεμελιωθεί και νομίζω πως θα, ήταν, θα είχε νόημα και άλλα εθνικά κοινοβούλια να ακολουθήσουν αυτή την οδό, ώστε κάποια στιγμή να μην ε, χρειάζεται πλέον καν να εξετάζεται, να, να, να δείχνουν ακριβώ την κάρτα σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα, όταν θα μπορούν μέσω συνεργασία με τι κυβερνήσει του να παρακολουθούν το τι ακριβώ συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε. Πρόεδρε, λέει ο κύριο Γκέρνη. Οι εθνικοί βουλευτέ που ξέρουν την λειτουργία και τη διαδικασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ε, ε, ε, θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Όχι, δεν λέω να υπάρξει σύγχυση αρμοδιοτήτων και έχει δίκιο η κυρία Μπερέ ότι θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, αυτή τη σύγχυση αρμοδιοτήτων. Να υπάρξει ενιαίο και διακριτό θεσμικό πλαίσιο για όλες τις πολιτικές και την εξωτερική πολιτική. Πάντως υπάρχει έδαφος και περιθώριο διερεύνησης του τι μπορούμε να κάνουμε. Α, και, και οι κάρτες κάτι λένε. Συνενώσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τι να σα πω, που μέχρι στιγμή οι συναντήσει μα με τα Εθνικά Κοινοβούλια έρχονται και επίτροποι να μιλήσουν και φέρνει, το φέρνουν τόση υπνηλία που θα έπρεπε να έχει βρεθεί ένα φάρμακο από τη βιομηχανία για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βαρεμάρα. Άρα Υπάρχει επομένω πολλέ φορέ ξύλινη γλώσσα, υπάρχει φλιαρία. Τέλο πάντων όλα κινούνται σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όλοι φεύγουν απογοητευμένοι από τέτοιε συναντήσει. Γιατί όλοι θεωρούν ότι αισθάνονται μια ματέωση τέλο πάντων όσον αφορά το ρόλο του. Τι να πει κοινοβουλευτικό νομοθεσία, έλεγχο εκτελεστική εξουσία, χάρη συμβολή στην πολιτική. Ε, τίποτα από αυτά δεν κάνουμε. Επομένω, πού είναι η σύνθεση που έπρεπε να προκύψει από τέτοιε συναντήσει. Οπότε πάμε εκεί να μιλήσουμε και τελικά μιλάμε δύο λεπτά ή ένα λεπτό. Να, υπάρχει περιθώριο διορθώσεων επομένω. Πάντως, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε τις εθνικές πολιτικές, έχουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές που είναι πέραν του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Να, έχουμε πούμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ανήκει στα 28 κράτη-μέλη και η διαχείρισή του απόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενεργεί ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Καμία ανάμειξη, κανένα δικαίωμα επ' αυτών από βάση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη βάζουν τον οβολό του για το ταμείο αυτό. Άρα, όποτε τα συζητάμε, τζάμπα κουβέντες είναι. Αν ρωτήσετε έναν εθνικό βουλευτή σχετικά, α, έχουν κάνει κάποια συνάντηση, μία και μόνη, όσον αφορά τον έλεγχο επί του Ταμείου. Σε σχέση με το δικό τους προϋπολογισμό, με τη δική τους κυβέρνηση που κάποια στιγμή βάζει τον οβολό στο Ταμείο. Και αρνητικά θα τοποθετηθούν οι εθνικοί βουλευτές. Και, για ρωτήστε. Ποιο κοινοβούλιο ασκεί περισσότερη επιρροή της Μπουρκίνα Φάτσο, Φάσο ή το Εθνικό Κοινοβούλιο στο οποίο τυχόν θα ρωτούσε κανένας τι γίνεται. Έχουμε και κάποιες κοινέ αρμοδιότητες και αφού πρόκειται για κάποιες κοινέ αρμοδιότητες τι να σας πω. Ε, θα πρέπει επίσης να οργανωθεί ο κοινό έλεγχος. Έχουμε συγκητές, έχουμε προέδρους επιτροπών που θα πρέπει να έρθουν σε επαφή και να συνοηθούν με τα εθνικά κοινοβούλια. Να ξεκαθαριστεί ποιο κάνει τι. Να κάτσω να κάνω μια καταγραφή του τι έχει γίνει. Να εξεταστεί πού υπάρχουν κενά στη διαδικασία του ελέγχου. Να, μια ιδέα. Άλλο. Πάντα μιλάω για την αναπτυξιακή μας πολιτική. Υπάρχει συνένεση στην Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη. Έχουμε κάποιες αρχές σχετικά. Έχουμε κάποιες δεσμεύσεις και στόχους. Ποσοτικά υπολογισμένους. Το 2005 ας πούμε είχαμε το σχετικό έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Συνένεση. Το προσυπέρεψαν τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Έτσι δεσμεύτηκαν οι 28 να δώσουν 0,7% ξέρω εγώ μέχρι το 2030. Εδώ και χρόνια και εγώ και άλλοι αναρωτιόμαστε. Γιατί να μην έχουμε περισσότερο έλεγχο και αξιολόγηση για, τις, ε, για τους στόχους. Δεν ασχολούνται τα κράτη-μέλη. Για πήγαινε να ρωτήσετε έναν υπουργό κάποιο κράτους μέλους όπως κάνει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Επιτροπή η Οικονομική να τον φωνάξουμε λοιπόν να έρθει εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξη και να εξηγήσει τι γίνεται σχετικά στη χώρα του. Θα αντιμετωπίσει κανεί αν το πει αυτό παχυλία διαφορία. Ε, αυτό είναι καρνάβαλο Ας σοβαρευτούμε. Αλλά όμω ούτε τα εθνικά κοινοβούλια έχουν το θάρρο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Να αναλύσουν τα τροτά του συστήματο, Να βρουν τα κενά. Να χαράξουν μια στρατηγική για να έρθουν αυτά τα κενά. Άρα στην επόμενη συνάντηση Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν δεν θυγεί αυτό το πρόβλημα ε, τότε θα είμαστε λάθος. Συνολικά. Επίσης έχουμε αυτόν τον ε, στόχο της 15 ετίας. Για το 2015 δεν είχε επιρρευθεί ο στόχος. Και λέμε θα πάμε για το 2030 και το 2028 που θα γίνει η επόμενη διάσκεψη για την χρηματοδότηση θα πει η Κομισιόν τι θα πει θα πει πάμε το 2045 μια που δεν πετύχαμε το στόχο ε, αυτό τι μας κάνει μας απλούς αδύναμους θεατές σε αυτό το γκαρνάβαλο νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερο. η Πρόεδρος σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση χρονοδιάγραμμα από τις εθνικέ ιδέες πρωτοβουλία είναι τα πράγματα πιο χαλαρά οπότε και θα έχουμε ένα εργαστήρι και καθόλου ελπίζω ότι τον Φεβρουάριο θα μπορέσουμε να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τον έγγραφο εργασία και κατόπιν ε, τον Μάρτιο θα γίνει συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, αυτά που είπες ε, Ζόρζ και τελική ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο του κειμένου τον Απρίλιο και ψήφιση τον Ιούνιο. Σας υπενθυμίζω ότι η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας έχει άλλου είδους δομή. Οπότε έχουμε την διευκρινιστική δήλωση και θα έχουμε την παρουσίαση των διαφόρων στοιχείων από τον εισηγητή. Τις συστάσεις, τις προτάσεις τις δικές σας μετά. να θέλετε και στη συλλογή των στοιχείων πραγματικών περιστατικών να συμβάλλετε και αυτό μπορείτε να το κάνετε σε συνεννόηση με τον Παύλο Δική του είναι έκθεση. Αλλά αν έχετε κάτι να συμβάλλετε μπορείτε να το κάνετε να πάρετε να τον βρείτε τον Παύλο Ωραία τέρμα με αυτό το σημείο στη μέση διάταξη. Τζορτζ, τι θα κάνουμε με το θέμα Πρέντα. Όλο το έργο είναι στην Ρωμανία, άρα δεν είναι εδώ ο Πρέντα. Α, να αρχίσουμε τώρα. Μπορείς εσύ να το πεις, ωραία, έκθεση Λίμπε. Όσον αφορά το θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση 2015. Thank you indeed. Yes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, νιώθω λίγο μόνος εδώ στα έδρανα του ΕΛΚ, αλλά όπως είπατε πολύ σωστά, ε, όλοι βρίσκονται σε συνάντηση του Προεδρείου ε, στο Βουκουρέστι. Ε, Σα διαβάζω λοιπόν τι παρατηρήσει του κυρίου Πρέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να παρευρεθώ ίδιος στην Επίτροπη για την συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σοφλίν που με αντικατέστησε. Η γνωμοδότηση τονίζει σημαντικές πτυχές που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκών, Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015. Καταρχάς, ε, ζητεί καλύτερη ε, εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν απαραίτητα μέτρα για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και του ευρέω κοινού. Επίσης, ε, θέλουμε πλήρη σεβασμό του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ε, της νομοθετικής και επίσης θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και κατά την συνεργασία μεταξύ των θεσμών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, καλούμε την ε, Επιτροπή ε, για να καθορίσει τα απαραίτητα βήματα για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, θέλουμε ενίσχυση του κράτους δικαίου. Οι δύο διάλογοι για το κράτος δικαίου από πλευράς του Συμβουλίου τονίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την καλύτερη λειτουργία του κράτους δικαίου. Δεν ε, έχω στόχο να ξεκινήσω συζήτηση σχετικά για μηχανισμό ε, δημοκρατίας, ε, κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συζήτηση στην ΛΥΜΠΕ συνεχίζεται. Άλλωστε νομίζω ότι η ΛΥΜΠΕ θα ε, ψηφίσει την Δευτέρα. Ο κύριος Πέραντα λοιπόν συνεχίζει ότι θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών και ελπίζω να έχουμε καλή και επιτυχή συνεργασία. Ευχαριστώ η Σίλβια Ιβον Κάουφμαν από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Νομίζω ότι έχει διατυπώσει τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε η Επιτροπή μας να διατυπώσει μια τέτοια γνωμοδότηση. Από τη δική μας πλευρά δεν νομίζω ότι απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις. Θα ήθελα στο σημείο 5... εκεί που μιλάει για ε, τον μηχανισμό ενίσχυσης ε, του κράτους ε, δικαίου. Έχουμε υιοθετήσει δύο ψηφίσματα με ευρεία πλειοψηφία και βρίσκω την ε, διατύπωση σημειώνει στο σημείο 5 πολύ ε, ασθενή. Επίσης ε, η ψηφοφορία στην ΛΥΜΠΕ για ε, την ενεργοποίηση μηχανισμού. Πιστεύω ότι αποτελεί, για το κράτο δικαίου πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου μας. Και επίσης ο χάρτης θεμελιωτών δικαιωμάτων ε, και το άρθρο 2 της συνθήκης θα πρέπει να αποτελούν ε, νομική βάση για νομοθεσία. Και επίση θα πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, νομίζω ότι... Ε, θα είναι ε, σημαντικό να έχουμε ευρεία πλειοψηφία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Morten... Ευχαριστώ. Μόρτεν Μέσσερ θέλει να πάρει το λόγο, όχι. Υπάρχει κανείς άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Εάν όχι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 11 Οκτωβρίου ή στις 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο θέμα της πρωινής μας συνεδρίασης. Ε, θα τα ξαναπούμε στις 2 και 4 με τους συντονιστές ε, στην ίδια αίθουσα και κατόπιν στις 3 ε, έχουμε την ε, συζήτηση με εμπειρογνώμονες. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε, διότι νομίζω ότι είναι μία από τις ε, πιο σημαντικές ε, συζητήσεις μας αφορά το Brexit. Θα σας δω λοιπόν το απόγευμα. Ευχαριστώ.